Otwieram posiedzenie. Άρχεται η συνεδρίαση. <clears throat> Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την προεδρία του απερχομένου Προέδρου του Κοινοβουλίου δεν πρόκειται να γίνει καμία συζήτηση. Δεν επιτρέπεται να συζητηθεί τίποτα που δεν αφορά την εκλογή του Προέδρου ή τουλάχιστον την επιβεβαιώση των εντολών. Δεν θα δεχτώ καμία παρατήρηση, καμία συζήτηση αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνον και αποκλειστικά με την εκλογή του Προέδρου, σύμφωνα με τον κανονισμό μας. Βάσει του κανονισμού πάντα, Είμαστε υποχρεωμένοι, σύμφωνα με το 13, να οργανώσουμε την εκλογή του Προέδρου. Το άρθρο 13 προβλέπει οι υποψήφοι να έχουν οριστεί από πολιτικές ομάδες ή τουλάχιστον από 40 βουλευτές. Και βάσει αυτών έχουμε λάβει τις τρεις εξής υποψηφιότητες που σας τις παρουσίασα και χτες αλλά θα σας τις ξαναπαρουσιάσω. Ο κύριος Νίτσιντεβα. Παρακαλώ, μπορείτε να σηκωθείτε να σας δούμε, κύριε Ντέβα. Μάρτιν, Παν Μάρτιν Σούλτς, πρόσε. Ο κύριος Μάρτιν Σούλτς. Παρακαλώ, κύριε Σούλτς. Η πάνη Νταϊάννα και η κυρία Ταϊάννα Βόλης. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω την παρατήρηση ότι με ειδοποίησαν οι υποψήφοι ότι είναι σύμφωνοι με την υποψηφιότητά της. Σας παρακαλώ τώρα μην σηκωθείτε πρόωρα από σας, γιατί θα σας ε, παρουσιάσω διάφορες οδηγίες στα πολωνικά. Εάν σηκωθείτε λοιπόν από τη θέση σας και δεν φοράτε πια ακουστικά, ίσως δεν θα καταλάβετε αυτά που έχω να σας πω. Βάσει του άρθρου 14, παράγραφος 1 του κανονισμού, ο υποψήφιος εκλέγεται ο... Εκείνος υποψήφιος εκλέγεται που έχει την πλειοψηφία των <laughs> εγκύρων ψήφων. Ε, Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια δεν θεωρούνται έγκυρη ψήφι. ποσου. Κατόπιν θα ήθελα να ορίσω διαψήφου οκτώ συναδέλφους που θα ασκήσουν το αξίωμα των ψηφολεκτών. εκλέγονται από το σύνολο των βουλευτών με κλήρο. Αυτή εδώ είναι η... Ε, εδώ έχω τα ονόματα των βουλευτών. Θα βγάλω τα, τα ψηφιακά. Είχα, έχω ένα όνομα. Πορσελίνο. Ε, κυρία, συμφωνείτε, κυρία Μπορσελίνο, συμφωνείτε να είσαστε ψηφολέκτης. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πρώτος ψηφολέκτης. Σόγκορ. Σόγκορ. Σόγκορ. Please stand up. Παρακαλώ σηκωθείτε να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε. Ωραία. The next. Επόμενος. Stiller. Lady or oh, lady or oh. lady. Madame Stiller. Α, η κυρία Στίλερ. Πού είναι, πού είσαστε. Συμφωνείτε. Όχι. Σας παρακαλώ, όχι, όχι. Συμφωνείτε, λέει ο πρόεδρος. Α, όχι, δεν κατάλαβα. Sorry, sorry. Congratulations. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για το μωρό σας, <laughs> κύριε Στήλερ. Great. So we will vote uh, Λοιπόν, αναπληρωτή. Αντί εσά. Πολύ ωραία. Παναγιώτοφ. Παναγιώτοφ. Do you agree? Συμφωνείτε? Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο. Green group, Where is Green Group? Not here. Απουσιάζει. Να βρούμε κάποιον άλλο τότε. Pots. Pots. Do you agree? Συμφωνείτε? Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Next is uh, Boris. Επόμενος Boris. Do you agree? Συμφωνείτε? Όχι? Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή έχω να υποδεχτώ μια αντιπροσωπεία της καζακικής ε, αντιπολίτευσης και πρέπει να είμαι στις δύο εκεί. Ε, it's a Να πάρουμε κάποιον άλλο, πάντο. Do you agree? Συμφωνείτε? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος. Καλινόφσκι. Do you agree? Συμφωνείτε? Ωραία. Θαυμάσια. Επόμενος. Καλφίν. Do you agree? Συμφωνείτε? Ευχαριστώ πολύ. And uh, the last one. Τελευταίος. Περέλο Ροντρίγκες. Where is he? Where is he? Do agree? Great. Συμφωνείτε? Θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας εξηγήσω τα επόμενα σημεία. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους βουλευτές που εξελέγησαν ως ψηφολέκτες να έρθουν εδώ και να κάτσουν πίσω από το Προεδρείο εδώ. Οι οκτώ αυτοί συνάδελφοι παρακαλώ να περάσουμε στη σειρά με την οποία εξελέγησαν. Ούρνη, αβιενς, παν, μπορσελίνο. Για να μπορέσει ο καθένας να είναι υπεύθυνος για μια κάλπη. Μπορσελίνο αλφαβήτα, Σόγκορ, ΣΕ, ε. Παναγιώτοφ, εφ έως Άσο, Πότς, Ιώτα Κάπα, Μπάγκο, Ελ ως Μ, Καλινόφσκι, Εν ως Έρα και Καλφίν, Εσ, Περέιο Ροντρίγες, Τε ως Αυτές είναι οι κάλπες για τις οποίες είναι εκάστοτε υπεύθυνοι συνάδελφοι. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι να έρθουν εδώ μπροστά και να ε, έρθουν εδώ πίσω από τα πέζια του Προεδρείου και να είναι εδώ κοντά μου. Just now, just now please. If you could come and to stand up behind me. Παρακαλώ τους ε, συναδέλφους ψηφολέκτες να έρθουν εδώ προς το Προεδρείο. Λοιπόν, δύο συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να έρθετε εδώ, πίσω από εμένα, στο Προεδρείο. Βλέπω έξι συναδέλφους συμφολέκτες εδώ, αλλά δύο συνάδελφοι ακόμη δεν έχουν έλθει. Proszę Państwa, So? Proszę Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πω συγκεκριμένα τώρα πώς θα ψηφίσετε. Ήδη έχετε πάρει τις οδηγίες ε, στο email, αλλά Ίσως δεν είχατε όλοι χρόνο να δεις διαβάσετε, γι' αυτό θα τις επαναλάβω. Πρώτα απ' όλα, θα σας διανεμηθούν τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι. Λοιπόν, αρχίσουν η διανομή των ψηφοδελτίων και των φακέλων. Παρακαλώ, να δοθούν σε όλα τα μέλη. Ακούτε όμως και τις οδηγίες που έχω να σας δώσω. Όσον αφορά την ψηφοφορία, θα ήθελα ακόμη μια φορά να σας υπενθυμίσω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Επαναλαμβάνω, απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Όταν πάρετε στα χέρια σας, λοιπόν, τα ψηφοδέλτια, θα πρέπει να γράψετε το όνομα του υποψηφίου τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε. Συγγνώμη, θα πρέπει να βάλετε σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε. Μην βάλετε δύο σταυρουδάκια, διότι θα είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο. Σταυρουδάκι, λοιπόν, δίπλα στο όνομα του υποψηφίου που θέλετε να ψηφίσετε. Εάν κάνετε λάθος, θα πρέπει να ζητήσετε από, τους, ε, από τα άτομα που σας δίνουν τα ψηφοδέλτια να σας δώσουν ένα άλλο ψηφοδέλτιο, ώστε με σαφήνεια να βάλετε στο βρός το όνομα του υποψηφίου που θέλετε να ψηφίσετε. Παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι να παραμείνετε στις θέσεις σας για να διεξαχθεί η ψηφοφορία. Δεν έχει αρχίσει ακόμη η ψηφοφορία. Λοιπόν, θα πρέπει τα ονόματα των συμμετεχόντων στην, ε, ε, στην εκλογική αυτή διαδικασία να υπάρχουν στα πρακτικά και γι' αυτό σας παρακαλώ να υπογράφετε τους καταλόγους που υπάρχουν δίπλα στην κάλπη. <clears throat> Επίσης θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχετε κάποιο έγγραφο στα χέρια σας για να αποδείξετε την ταυτότητά σας. θα βάλει τα ψηφοδέλτια στο φάκελο αφού τα διπλώσετε και θα βάλετε τον φάκελο στην κάλπη. Είπαμε μόνο ένα σταυρό, όχι δύο και όχι σχόλια. Υπάρχει ένα θέμα για την ε, διαδικασία την εκλογική, κύριε Σλούτερ. Μάλιστα, πρόεδρε, σύμφωνα με τις διαδικασίες, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει, επί και, να έχει υποβάλει επίκαιρα στοιχεία για τα οικονομικά του συμφέροντα. Το έχουν κάνει αυτό όλοι οι υποψήφοι. Ε, ναι, ναι. Έχουν όλα διακανονιστεί και διευκρινιστεί και εξεταστεί βάσει των νέων κώδικα και υπάρχουν τρει μήνες προθεσμία για να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ να πάτε στην ε, κάλπη με τα αρχικά του ονόματό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 Συμβολικά. Συμβολικά. Όχι, εστιανέ, που για κάθε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

Dear friends, I will check. Αγαπητοί φίλοι, θα ελέγξω τώρα κατά πόσον ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Η κυρία Βαρσελίνο, α ως β. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία σε εσά. Madame Borsellino, our colleague, box A, B, have you finished? Στο, στην κάλπη ΑΒ τελειώσατε με την ψηφοφορία ή ακόμα. Okay, you are coming. Okay. Uh, ολοκληρώθηκε, έρχεστε. Εντάξει. Κάλπη C έως C. Κύριε Σόγκο, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ναι. Ωραία λοιπόν. Κάλπη FJ. Κύριε Παναγιώτοφ, ολοκληρώσατε την ψηφοφορία. Κύριε Παναγιώτοφ, ολοκληρώσατε. Not yet. Okay. I will... Όχι ακόμα, ωραία, θα περιμένω. Okay. I will wait. Θα περιμένουμε λοιπόν. Mrs. Great, great. We will wait. Box A, B is coming to me. Η κάλπη AB έρχεται. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ο κύριος Πολ, συνάδελφος, για την κάλπη LM ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάγκο. N έως R, ολοκληρώσατε. Είστε έτοιμος. Ωραία. Ο κύριε Καλινόφσκι. Το S. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Τελειώσατε. Okay. Κάλφιν, ε, S. Κύριε Κάλφιν, το S ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έχουμε έξι άτομα που δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Και το ο Z. κύριε Περέρο Ροντρίγες, ολοκληρώσατε τη διαδικασία. Ωραία. Εξαιρετικά. Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να ψηφίσει. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ψήφισαν όλοι. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, αγαπητοί συναδελφοί, ο... κλείνω εδώ τη διαδικασία της ψηφοφορίας και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους ψηφολέξεις να πάνε στην αίθουσα R01-101 για να κάνουν την καταμέτρηση και διακόπτεται να μεταξύ η συνεδρίαση. Και θα συνεχίσει η συνεδρίαση όταν χτυπήσει το κουδουνάκι και θα υπάρχει και αναγγελία και στις οθόνες. Σε 30-40 λεπτά θα ακούσετε το κουδούνι και θα πρέπει να ξανάρχετε εδώ στην Ολομέλεια. 40 λεπτά περίπου υπολογίζω. Διακοπή λοιπόν της συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ.